Mr. Ich habe für diesen Bericht gestimmt. Τοποθετήθηκα έτσι ψηφίζοντα υπέρ τη ασφάλεια των παιδιών. Διότι ζητείται μια μεταρρύθμιση σε σχέση με πρόσθετα μέτρα για ασφαλή διαβατήρια ή βιομετρικά στοιχεία. Ε, συνολικά ένα πακέτο λοιπόν το οποίο μα οδηγεί προ τα εμπρό στην καταπολέμηση τη εμπορία παιδιών και για την αύξηση της ασφάλειας υπέρ των παιδιών. Ευχαριστώ Ευχαριστούμε. Η κυρία Ρόιτοβα. Για η ασφάλεια των διαβατηρίων πρέπει να ενισχυθεί με τα βιομετρικά στοιχεία. Αυτό είναι καλό για την ασφάλεια των Ευρωπαίων Πρέπει όμως να δούμε και την αντίθετη πλευρά. Πώς θα προστατευτεί η ιδιωτική ζωή. Θα πρέπει να εφαρμοστεί νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο χωρίς γραφειοκρατικούς φραγμούς ή κατάχρηση των πληροφοριών. Η Ευρωπόλ και το Frontex πρέπει να συνεργάζονται σε αστυνομικό επίπεδο για να υπάρξει περισσότερη ασφάλεια στην Ευρώπη. Είναι καλό που θα έχουν διαβατήριο και οι δωδεκαετής γιατί αυτό θα αποτελέσει καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Ευχαριστούμε Βάνεκ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Στα νέα διαβατήρια, για τα νέα διαβατήρια υποστήριξα την έκθεση Κοέλιο γιατί νομίζω ότι είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και την καταπολέμηση της πλαστογράφησης των διαβατηρίων. Πρέπει στις χώρες Σέγγεν να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα για να υπάρχει εγγύηση του ανοίγματο των συνόρων έτσι ώστε να προστατεύονται οι τίμοι και να καταπολεμούνται οι άτιμοι. Αλλά τα καλύτερα αυτά διαβατήρια δεν είναι ιδεώδης λύση γιατί κάθε φορά εκατοντάδες χιλιάδες παράνομοι μετανάστες εισέρχονται στην Ευρώπη καθώς και ήμοι παράνομοι. Στη χώρα μου το Βέλγιο δηλαδή 77.000 ζήτησαν νομίμως μετανάστευση και ακόμα μεγαλύτερος αριθμός εισήλθε παρανόμως. Επομένως δεν είναι πανάκια τα βιομετρικά αυτά διαβατήρια. Ο κύριος Στογιάννοφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ καταψήφισα την έκθεση Κοέλιο για δύο λόγους. Πρώτον, Ανησυχώ για τις πολιτικές ελευθερίες. Τα βιομετρικά στοιχεία απειλούν την ασφάλεια των πολιτών, την ελευθερία τους. Και τίθενται κατά, είναι κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ελευθερία της μετακίνησης, παραδείγματος χάρη η χορήγηση αυτών των διαβατηρίων θα αλλάξει διαδικασία για δεύτερη φορά σε πολύ λίγο χρονικό, μικρό χρονικό διάστημα στη χώρα μου. Και τα χρήματα που απαιτούνται για την αγορά αυτών των διαβατηρίων είναι πάρα πολλά. Είναι ακριβό. Και αποτελεί πρόσθετο βάρος για τους ηλικιωμένους ιδιαίτερα η απόκτηση αυτών των διαβατηρίων 50 ευρώ. Γι' αυτό καταψήφισα. Μίτσελ. Ευχαριστώ. Εγώ καταψήφισα την έκθεση Καπάτο γιατί πιστεύω ότι υπάρχει μια καλύτερη έκθεση για τα ίδια θέματα. Επίσης όμως το Κοινοβούλιο πρέπει να κάνει κάτι ως προς τα πρακτικά του και τα αρχεία του. Υπάρχουν εδώ παρόντες βουλευτές επί 4,5 χρόνια και μιλούν πάρα πολύ λίγο. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Μερικοί δεν συμμετέχουν στη δουλειά του Κοινοβουλίου, ούτε στην Ολομέλεια, ούτε στις Επιτροπές. Και μετά έρχονται εδώ πέρα και μιλάνε. και περνάνε του, όλο τους το χρόνο στα κράτη-μέλη και όχι εδώ. Μα η δημοκρατία πώς θα εφαρμοστεί αν οι ευρωβουλευτές πληρώνονται αλλά δεν προσέρχονται. Αυτό είναι κατάχρηση της δημοκρατίας και πρέπει να το τονίσω. Όταν ζητάμε περισσότερη διαφάνεια τότε πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχουν και ορισμένοι βουλευτές που δεν κάνουν τη δουλειά τους. Κύριε Μίτσελ, στην ουσία εσείς κάνατε επεξήγηση ψήφου για την έκθεση Καπάτο, ενώ μιλούσαμε για την Κοέλιο. Δεν θα σας δώσω το λόγο για την έκθεση Καπάτο. Προχωράμε στην έκθεση Λάμστορφ και έχουμε ένα αίτημα για επεξήγηση ψήφου από την κυρία Ροϊτόβα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Η αγορά αγαθών είναι κατακαιρματισμένη και δυσλειτουργική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ανοιχτεί αυτή η αγορά όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες και λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 3 της συνθήκης κατέβαλα κάθε προσπάθεια στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή να τερματιστεί η διασπάθηση δημοσίων κονδυλίων η εθνική νομοθεσία σε σχέση με την εφαρμογή για τις ε, κρατικές προμήθειες ε, στρατιωτικού υλικού που δεν έχουν καμιά σχέση με την ε, διαφάνεια. Η παρούσα πρόταση θα εξοικονομήσει χρήματα και θα μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει υπέρ της χρήσιμης τεχνολογίας οπλικών συστήματων. Thank you, President. opposed report εγώ κατεψήφισα διότι νομίζω ότι υπάρχει ένας κίνδυνος για τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις που επενέβησαν τόσο πολύ για την άμυνα και τώρα δεν έχουν κέρδη. Δεν έχουν. Διότι σύμφωνα με την προτινόμενη αυτή οδηγία χρειάζεται να ανοίξει στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό λέει η προμήθεια ακόμη και για χώρες που δεν μπορούν να προστατεύσουν τις χώρες εργασίας και στο Ηνωμένο Βασίλειο ιδιαίτερα τίθεται αυτός ο κίνδυνος. Ανησυχώ ιδιαίτερα γιατί θέλω να υπάρξει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ασφάλεια στα πλαίσια της ΚΕΠΑΣ μάλλον παρά να αυξάνονται με μονομένα ατομικά κέρδη. Ο κύριος Φατούτσος. Δεν το θέλει αυτό. Ευχαριστώ. το διακεκριμένο κοινό που με ακούει. Εγώ ζήτησα το λόγο μόνο για να πω ότι ψήφισα υπέρ της έκθεσης Λάμσδορφ που κινείται ένα βήμα μπροστά για την κοινή άμυνα και ασφάλεια αλλά διερωτώ πότε επιτέλους θα έχουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή άμυνα ένα πραγματικό ευρωπαϊκό στράτο, ένα, μια πραγματική δυνατότητα να εξοικονομήσουμε χρήμα και να μπορούμε και να υπερασπιστούμε την Ευρώπη ως Ευρώπη. Ελπίζω, Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ. Ε, εδώ δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση, θα ήταν εξαιρετικά περίπλοκο. Ε, ε, προχωράμε στις επεξηγήσεις ψήφου για την έκθεση Σλίτερ και ζήτησε το λόγο η κυρία Ροϊτόβα. Σας ευχαριστώ για την πρόταση για τις επικίνδυνες ε, ουσίες που την υποστήριξα επειδή η προσπάθεια είναι το χλωρομεθάνιο για τις ε, διάφορες διαλύσεις να χρησιμοποιείται για τα διάφορα διαλύματα υπό περιοριστικούς όρους ε, και με αυστηρούς όρους. Είμαι επισμένη ότι αυτές οι εξαιρέσεις ε, δεν θα χρησιμοποιηθούν καν διότι υπάρχουν ήδη εναλλακτικέ λύσεις όχι μόνο για τους καταναλωτές αλλά και τους επαγγελματίες. Κυρία Σίνοτ, έχετε το λόγο. Ορισμένες ουσίες είναι τόσο επικίνδυνες που θα πρέπει τελείως να απαγορευτούν. Εν πάση περιπτώσει να περιοριστεί η χρήση τους πολύ αυστηρά από εξαιρετικά αυστηρού ε, και νόμους υγείας και ασφάλεια. Αυτή είναι μια από αυτέ τι ουσίες και πρέπει να βγει από την κυκλοφορία. Σα ευχαριστώ και τώρα προχωράμε στην έκθεση Φιγκερέντο. Ζήτησε το λόγο η κυρία Ρόιτοβα. Θα ήθελα να αναφερθώ ότι σε σχέση με τους όρους εργασίας ε, για τον, τομέα, τον επαγγελματικό για την αλληλεία, διότι οι αλληλείς έχουν δικαίωμα να έχουν ε, θετικές ε, προϋποθέσεις, όρους απασχόλησης. Υπάρχουν πολλά τυχήματα. Το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να ζητηθεί να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε ταχύτερα να εφαρμοστούν αυτές οι αρχές πριν από το 2012. Γι' αυτό τοποθετήθηκα σε αυτή την έκθεση με αυτόν τον Έχουμε τώρα δηλώσει επεξηγή ψήφου για την έκθεση Κατάνια. Ε, παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο σα, γιατί είσαστε πολλοί που θέλετε να μιλήσετε. Πρώτα, η κυρία Μπελοχόρσκα. Η έκθεση πρωτοβουλία του Κατάνια προκάλεσε μεγάλη αντιπαράθεση απόψεων ανάμεσα στου ευρωβουλευτέ. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε να κάνουμε ταυτόχρονα με πολύ σοβαρά προβλήματα, οικονομική και ενεργειακή κρίση, ε, σύγκρουση ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρωσία και ακριβώ αυτή τη στιγμή πρέπει να ενεργήσουμε ενωμένα και να ε, περιορίσουμε τι απειλέ στα σύνορά μα. Η κρίση αφορά όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπληξε τους Σλοβάκους, τους Ούγγρους, τους Γερμανούς κτλ είναι προβλήματα τα οποία επανέρχονται με κάποια περιοδικότητα στο κοινοβούλιο μας. Δεν μπορούμε αυτό να το αγνοήσουμε. Πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή στην επίλυση προβλημάτων, στην εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης. Επανειλημμένος εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Έχουμε πει πως η αυτονομία στο πλαίσιο του κοινού μας ευρωπαϊκού χώρου δεν σημαίνει ε, αποδοχή. Η βασική ιδέα της διεύρυνσης της Ένωσης δεν μπορεί να αγνοηθεί, να απορριφθεί. Πρέπει να θυμόμαστε αυτά που έλεγε ο Σούμαν. Δηλαδή, ένας Ευρωπαίος που σκεπτόμενος δεν μπορεί να είναι ευτυχής για την δυστυχία του γειτονά του, γιατί όλοι ναι. έχουμε κοινό, κοινή μοίρα για το καλό ή για το κακό. Um Για την έκθεση Κατάνια. Αυτή η έκθεση είναι πραγματικά ένα μεγάλο πακέτο χωρίς δυνατότητες ελέγχου πώς τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2004 στο 2008 τηρήθηκαν. Είναι απλά μια παρήθμιση ως κατάλογος των πολιτικά αριστερόστροφων και μεταξύ άλλων και την ε, αναγνώριση της ισότιμης λέει σεξουαλικής σχέσης ε, ομοφιλοφίλων, νομιμοποίηση ναρκωτικών, νομιμοποίηση ευθανασίας, ε, νομιμοποίηση κάθε παράνομης δράσης. Αυτή η απαρίθμηση που με πλειοψηφικό τρόπο υιοθετήθηκε από μένα, από την αντιπροσωπεία του ΕΛΚ συνολικά απορρίπτεται κάθετα. Και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πω ότι καταψηφίσαμε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Υπερψήφισα την έκθεση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ένωση 2004-2008. Αυτή η υποστήριξη προκύπτει από το γεγονός ότι δεν υιοθετήθηκε αρχική πρόταση για το άρθρο 49 δηλαδή για την ε, περιφερειακή και εδαφική αυτονομία. Είναι ένα όχι κάθαρο και σαφές απέναντι στους ε, συνομότους που θέλουν να ε, παίξουν με το στάτους που Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν δέχεται αυτά τα παιχνιδάκια για την τοπική και ταφική αυτονομία. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ όλους όσους ενέκριναν αυτό το αποτέλεσμα. Κυρία Ροϊτόβα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, και εγώ καταψήφισα την έγκριση αυτής της έκθεσης του κομμουνιστή ευρωβουλευτή όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταψήφισα, γνωρίζω ότι τώρα μπορέσαμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα και αυτό είναι καλό για τις μειονότητες. Κάποια πράγματα όμως αντικειμενικά δεν είναι καλά και δεν βαίνουν καλώς. Διότι εδώ έχουμε μια χωρίς προηγούμενο υπέρβαση των αρμοδιοτήτων κατάχρηση αρμοδιοτήτων. Τα δικαιώματα αυτά μονομερώς ε, ερμηνεύονται πολιτικά και η αρχή της επικουρικότητας περιορίζεται και περικόπτεται και η δυνατότητα των κρατών μελών περιορίζεται. Εγώ ψήφισα κατά της έκθεσης Κατάνια κύριε Πρόεδρε Και είναι κρίμα που μια έκθεση που καλύπτει τόσα πολλά θέματα να περιλαμβάνει και ορισμένα που είναι εκτός των δικαιοδοσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ, εδώ το Γι' αυτό καταψήφισα, γι' αυτό. Στην Ευρωβουλή έστ, παιδιά, τι Δεν κοπείτε. Πολλέ από τις ε, ελλείψεις ε, σε σχέση με τις ε, πολιτικές μειονότητες, για τις μειονότητες έχουν απορριφθεί. Γι' αυτό και καταψήφισα την έκθεση στην Ουγγαρία. Έχουμε μειονότητες. Αυτή η έκθεση μιλά για προστασία των μειονοτήτων, αλλά και φυσικά ένα θεμελιώδες δικαίωμα είναι το δικαίωμα να μιλά κανείς τη γλώσσα του. Δεν μπορούν να το κάνουν όλες, αυτές, όλες οι μειονότητες αυτό μέχρι στιγμής. Στην Ευρώπη έχουμε 150 μειονότητε. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλήξουμε σε έναν ορισμό του τι εστί μειονότητα. Παράγραφο 49, την αυτοδιαχείριση και αυτοδιάθεση των μειονοτήτων. Νομίζω ότι είναι μια τέλεια διατύπωση για αυτό το στόχο. Οι βέλτιστε πρακτικέ πρέπει σχετικά να ακολουθούνται αυτές που υπάρχουν ε, και είναι διαθέσιμες. Βέλτικες, βέλτιστες πρακτικές. Thank you, President. A society consumed by rights is a... Μια κοινωνία που ζητάει όλο δικαιώματα και όλο να παίρνει έχει όρια. Και σε αυτό βασίζεται το αίτημα της έκθεσης για ισότητα μεταξύ κανονικών ζευγών και ομοφιλοφίλων δεσμών. Ο φυσικός νόμος είναι ένας άντρας και μια γυναίκα. Υπάρχει διαστροφή όταν ζητάμε ισότητα και για το αντίθετο. Όσο και να είναι της μόδας, ο ανατροσίμητρη, η φυσική πραγματικότητα η ίδια απαιτεί να μην τα εξισώσουμε. Το δικαίωμά μου να πάρω αυτή τη θέση είναι μικρότερο από το δικαίωμα των υπολείπων να ζητάνε την αντίθετη. Εγώ διαφωνώ με την έκθεση και αυτό τι με κάνει γελίο δεν με πειράζει γιατί είμαι υπέρ του σωστού και όχι του λάθους. Κύριος Βανέκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε σταδιοδρομία μου σε αυτή την Ευρωβουλή σπάνια τόσο μεγάλο κατάλογο μεγάλων ανοησιών είδα ποτέ μου και τέτοιων κοινοτοπιών όπως εδώ στην έκθεση Κατάνια. Σπάνιο αυτό ευχάριστο και ωραίο ότι σε μια έκθεση γίνεται λόγος για τα θεμελιώδη δικαιώματα και για γίνεται αναφορά στη συνθήκη της Λισαβόνας πέρα από δημοψηφίσματα και δεν υπάρχει καμιά νομική βάση για όλα αυτά και δεν υπάρχουν και εχέγγυα. Εχέγγυα υπάρχουν τα θεμελιώδη δικαιώματα για τους Ευρωπαίους πολίτες, ναι, αλλά εδώ φαίνεται για την ευρωκρατία να πρέπει να ισχύουν αυτά αποκλειστικά και πιστεύω ότι οι πολίτες από τη χώρα μου σίγουρα στην ίδια τη χώρα δεν μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς πια για την ευημερία τους, για τη γλώσσα τους, για τις παραδόσεις τους θα πρέπει να τις ε, υπερασπίζονται και να είναι και ευγνώμονες για το ότι μπορούν να τις υπερασπίζονται. Αυτό είναι μια ένδειξη της πολιτικής ορθότητας. Με την έκθεση Κατάνια γελιοποιήθηκε το Κοινοβούλιο για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και ο τρόπος πώς ασκείται αυτό το δικαίωμα χωρίς αμφιβολία είναι το πιο σημαντικό θερμόμετρο ή δείκτης για την κατάσταση των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στην έκθεση απευθύνεται προειδοποίηση για την αυτολογοκρισία που έγκυται στο ότι κάποια θέματα αποκλείονται από την κοινή συζήτηση ή από το επίκεντρο. Υπάρχουν ε, κάποια εδάφια στην έκθεση που γίνεται αναφορά σε άτομα σε ομάδες που ε, οδηγούνται στο να σιγούν ή να ε, αποσιωπούνται οι θέσεις τους και υφίστανται και επιθέσεις. Εκείνο όμως το οποίο είναι απαράδεκτο είναι η μεσθένος δίωξη των κηρυγμάτων μίσους και των άρθρων εκείνων όπου γίνεται ε, προπαγάνδα μυσαλλοδοξίας. Αυτό είναι ακριβώς το θέμα της αυτολογοκρισίας όπου αλλού σε, άλλα εδάφια αποτελεί αντικείμενο επικρίσεων και σε εμάς το μεγαλύτερο φλαμανδικό κόμμα καταδικάστηκε λόγω των παρεμβάσεών του για την μεταναστευτική πολιτική. Εδώ πώς μπορεί να τοποθετηθεί κανείς υπέρ της ελευθερίας έκφρασης. Ή είναι κανείς υπέρ της ελευθερίας έκφρασης με, όλες, με ό,τι συνεπάγεται αυτό ή είναι κατά κανείς. Ο κύριος Φαντούτσο. για τα θεμελιώδη δικαιώματα, αν και καταψήφισα στην τελική ψηφοφορία ήμουν υπέρ της παραγράφου 81. Ο φίλος μου λοιπόν Γιούστος Κατάνια το πρέπει να το ξέρει για να διευκολυνθούν εγώ είμαι υπέρ της διευκόλυνσης της πρόσβασης των νέων και των ηλικιωμένων και των αναπήρων στην αγορά εργασίας. Ο Κατάνια σωστά θεώρησε ότι η βελτίωση στην πρόσβαση στην εργασία σημαίνει και βελτίωση στην πρόσβαση σε συντάξεις. Γι' αυτό μίλησα για νέους ηλικιωμένους και αναπήρους και ξέρω ότι Σίγουρα θα συμφωνεί και ότι πριν φτάσει κανείς μέχρι τη σύνταξη ή μάλλον ότι οι νέοι αρχίζουν ως νέοι και καταλήγουν ως συνταξιούχοι. Αυτά τα λέω γιατί. Για να τονίσω ευπρεπώς ότι και οι ηλικιωμένοι έχουν δικαίωμα σε σύνταξη. Η κυρία σύνα. Σε αυτή την έκθεση κατάνοια ορισμένοι χρη... Χρησιμοποιούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα για να δικαιολογηθούν οι εκτρώσεις. Δεν είναι το σημαντικότερο από τα δικαιώματα αυτά το δικαίωμα στη ζωή, από το οποίο εξαρτώνται όλα τα υπόλοιπα. Και ως Ιρλανδί βουλευτής και ψηφοφόρος, θα ήθελα να τονίσω ότι η Χάρτα των Θεμελιωδών και η Συνθήκη της ε, Λισαβόνας η ίδια επίσης επικροτούν την έκτρωση. Η κυρία Μακ Γκίνες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα οι υπηρεσίες να γνωρίζουν ότι για την παράγραφο 31 είχα ψηφίσει υπέρ. Η έκθεση αυτή θα έπρεπε να λέει περισσότερα για τους αναπήρους. Παρ' όλα αυτά χαίρομαι που ενεκρίθη η τροπολογία 42 που ζητάει τα χρήματα να δίνονται μόνο στις χώρες που εφαρμόζουν αυτά που προβλέπει ο ΟΗΕ. Υπάρχουν πολλά θέματα στην έκθεση που θίγονται στην έκθεση που είναι όμως θέματα επικουρικότητας και όχι για την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δεν νομοθετεί ούτε πρέπει να νομοθετεί για θέματα όπως τις εκτρώσεις. Γι' αυτό απέσχον τελικά στη συνολική ψηφοφορία. Έσχος αν και με την τροπολογία που ανέφερα δίνεται λόγο σε εκείνους που δεν τον έχουν. Ο κύριος Μικολάτσικ. Στο πολύ. Η έκθεση Κατάνια αφορά βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Συμφωνώ με ορισμένους προλαλήσαντες και προλαλήσασες ότι τα κύρια στοιχεία της έκθεσης απορρίφθηκαν. Και αυτό διορθώνει την αρχική έκθεση. Γιατί τα λεγόμενα σεξουαλικά δικαιώματα συμπεριλαμβάνουν και το δικαίωμα στην έκτρωση. Αυτό επιβάλλεται τελικά στα κράτη-μέλη, χωρίς συζήτηση. Πρόσεξε. Εγώ είμαι υπέρ της προστασίας της ανθρώπινης ζωής από τη σύλληψη. Έμπενερ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Εγώ συμμερίζομαι τα όσα είπε εδώ ο κύριος Πίρκερ και γι' αυτό και δεν χρειάζεται να ε, καθυστερήσω. Πιστεύω πως ε, ο κύριος Κατάνια είναι εκτός θέματος. Η έκθεση αυτή δεν θα έπρεπε καν να έχει φτάσει εδώ στην Ολομέλεια, γιατί θα έπρεπε οι υπηρεσίες να επαληθεύσουν αν μία έκθεση ε, αναφέρεται στον τίτλο που φέρει ή αν είναι άλλον άλλον. Αυτή η έκθεση λοιπόν είναι τελείως εκτός θέματος και δεν αναφέρεται στον τίτλο της και στο θέμα της όσον αφορά ένα συγκεκριμένο θέμα, mm. εκείνο της παραγράφου 49, θα είχε... Θα προτιμούσε ε, το σώμα να έχει υιοθετήσει το αρχικό κείμενο, να μην το τροποποιήσει. Εγώ καταψήφισα την έκθεση στο σύνολό τη. Ακριβώς για τους προαναφερθέντες λόγους. Ευχαριστώ κύριος Δίλαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ σπάνια με τέτοια πεποίθηση και στένος καταψήφισε μια τέτοια έκθεση όπως αυτή σήμερα. Αν ακολουθήσουμε τις συστάσεις αυτής, αυτής της έκθεσης, τότε αύριο πού θα καταλήξουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχουμε μια δικτατορία της πολιτικής ορθότητας που θα έχει επιβληθεί. Υπό το πρόσχημα λέει της καταπολέμησης του ρατσισμού και υπό το πρόσχημα της υπεράσπιση της ελευθερίας της έκφρασης και όσον αφορά και θέματα μετανάστευση. Λοιπόν αυτή η έκθεση θέλει να ανοίξει πόρτα και παράθυρο στην παράνομη μετανάστευση ακόμα πιο πολύ από όσο έχει ανοίξει. Και εδώ δεν πρόκειται για δικαίωμα της ελευθερία των πολιτών και τη ασφαλεία του. Πρόκειται για δικαιώματα εγκληματιών Δικαιώματα και υποχρεώσεις όμως συνδέονται σε μια κανονική κοινωνία. Εδώ όμως δεν βλέπω σε αυτήν την έκθεση να γίνεται λόγος για οποιαδήποτε υποχρέωση των αλλοδαπών να σέβονται και να εντάσσονται στις αρχές της, ε, των κοινωνιών μας. Το αντίθετο, μέχρι κορεσμού δακτυλοδεικτούμε ως υπεύθυνου ε, τους ε, Ευρωπαίους και τους στιγματίζουμε. Φτάνει πια. Δεν είναι δυνατόν με αυτόν τον τρόπο να γίνεται κατάχρηση.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 Έκθεση Κατάνια. Πολλά από αυτά με βρίσκουν σύμφωνα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία, με τα οποία διαφωνώ. Α πούμε, δεν θεωρώ ότι είναι ζήτημα, ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασχολείται με τα δικαιώματα των πολιτών. Επίσης, ε, δεν δέχομαι τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, που είναι ένα πολιτικό κείμενο, το οποίο μαγειρεύτηκε ε, λόγω τη αποτυχία του Ευρωπαϊκού Συντάγματο σίγουρα δεν είναι βρετανικός, ε, ευρωπαϊκός νόμος και, και ακόμη πιο σίγουρα δεν είναι βρετανικός νόμος αυτό. Απορρίπτω τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είμαι κατά της, απόλυ... της απόλυτης προσέγγισης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης ε, κατά της αναγνώρισης ε, των ε, ζευγαριών του ίδιου φύλου, αλλά και πάλι δεν είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά των κρατών μελών. Γι' αυτό και καταψήφισα αυτή την έκθεση. Κύριε Πρόεδρε, η... πείρα μας διδάσκει ότι τα δικαιώματα αυτά στα χαρτιά δεν επαρκούν για την άσκησή τους. Τα δικαιώματα τα οποία αναφέρονται στη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών δεν είναι τόσο διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται για παράδειγμα στα συντάγματα της Ανατολικής Γερμανίας και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Όμως δεν ήταν ικανοποιημένοι οι πολίτες αυτοί με τέτοια δικαιώματα. Είναι άχρηστα τα τέτοια δικαιώματα στα χαρτιά χωρίς να υπάρχουν μηχανισμοί επιβολής τους. Ε, δεν είναι δυνατόν να, δεχθούμε μια τέτοια κρίση. Υπάρχει κρίση δημοκρατική νομιμότητας όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας τρόπος να βελτιωθεί αυτή η κρίση θα ήταν να είμαστε πιστοί στου ε, ψηφοφόρους μα και την συνθήκη τη Λισαβόνα ε, να την θέσουμε υποσυ σειρά ε, δημοψηφισμάτων να δούμε ποια θα είναι η έκβασή Σε Ευχαριστώ. Και Κυρία Τόμασεύσκα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει εδώ το δικαίωμα για τα παιδιά ο ιδίου φίλου, για, την, για γάμους ιδίου, ιδίου φίλου και για τα διαζύγια δεν θα πρέπει να είναι οι υπάλληλοι εκείνοι οι οποίοι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα αποφασίζουν τι θα γίνεται και τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ε, έρχονται σε επαφή και να μιλούν με τους γονείς τους ε, στη μητρική τους γλώσσα. Αν μιλούν διαφορετική γλώσσα οι γονείς πρέπει και τις δύο γλώσσες να έχουν στη διάθεσή τους. Όμως στην Γερμανία παιδιά μεικτών γάμων υφίστανται το πλήγμα του ότι δεν επιτρέπεται να μιλάνε πολωνικά με τον πολωνικό γονέ, πολωνό γονέα τους. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υποστήριξα την τροπολογία 24. Η απόρριψη όμως αυτής της πρότασης με οδήγησε στο να καταψηφίσω την έκθεση συνολικά. Επίσης θέλω να υπογραμμίσω το δικαίωμα στη ζωή που είναι σημαντικό και την αρχή της επικουρικότητας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάτεν παρακαλώ. Thank you, Mr. President. Ε, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Βρετανικό Κόμμα Ανεξαρτησίας είναι κατά του ρατσισμού, κατά του γυναικείου κοτριασμού, κατά των ε, προκαταλήψεων για την ε, ομοφιλοφιλία οπουδήποτε στον κόσμο. Ωστόσο, οι Βρετανοί χαίρουν ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και δεν χρειάζονται την προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μη δημοκρατική και αντιδημοκρατική και γι' αυτό και δεν αποτελεί τον κατάλληλο φύλακα οποιοδήποτε ανθρώπου όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Επίσης, οικογενειακό δίκαιο είναι θέμα των κρατών μελών και δεν είναι θέμα δικαιοδοσίας της Ένωσης. Τώρα, για το αν οι ε, τοξικομανείς θα πρέπει να ε, διώκονται ποινικά ή όχι θα είναι και πάλι θέμα κρατικό και δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντικαταστήσει τα, τα δικαστικά συστήματα των κατώμελων και γι' αυτό και καταψηφίσαμε την έκθεση αυτή. Ο κύριος Ήτον Χάρης, παρακαλώ, πρόεδρε. Θα έπρεπε όταν μιλάμε για τέτοιες εκθέσεις την συζητώ με εθελοντές και εκπροσώπους από τη δική μου εκλογική περιφέρεια. Μπορεί κανείς από τα βιώματα και με τέτοιου είδους επαφές να αποκομίσει πολλές γνώσεις και προσπαθώ και με άλλους ε, βουλευτές να συζητήσω και από άλλες πλευρές ε, του πολιτικού φάσματος να δω ποια είναι τα βιώματα και απόψεις άλλων. Συμφωνώ απόλυτα με τις απόψεις που εκφράστηκαν από, τον, από τους συναδέλφους Χάναν για παράδειγμα και σας θέματα για αυτή την έκθεση θα ήθελα να αναφερθώ στον κύριο Άλιστερ που δεν ήταν της δικής μου πολιτικής ομάδας ε, και που εργάστηκε σκληρά και που η σύμβουλή του είναι αξιολογική καθώς τον γνωρίζω σε σχέση με την συμφωνία να διαφωνήσω μαζί του, θα έπρεπε να το υπογραμμίσω αυτό. Μια έκθεση όπου με ευχολόγια μπορεί κανείς να ε, απαριθμίσει θέματα σε καταλόγους, ε, είναι εύκολο να ε, δεχθεί κανείς, είναι εύκολο να ακολουθήσει κανείς με τέτοια πορεία. Εγώ όμως απήχα, ευχαριστώ. Η κυρία Γκάλ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτή η έκθεση για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι είναι μια πολύ περίπλοκη σύνθετη έκθεση που είναι μια νέα απαρχή, ένα σημαντικό βήμα όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών και τα θεμελιώδη δικαιώματα στον κοινωνικό τομέα. Τα δικαιώματα των μειονοτήτων και η προστασία τους ε, ως ε, θέμα είναι κάτι που πρέπει να αξιολογήσουμε με πολύ θετικό τρόπο και όσον αφορά και την αυτονομία ή και την χρήση μιας γλώσσας από μια μειονότητα. Αυτά είναι θετικά. Υπερψήφισα λοιπόν εγώ και γι' αυτό η Ουγγρική Αντιπροσωπεία στο ΕΛΚΑ υπερψήφισε αυτή την έκθεση παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές παράγραφοι που από εμάς δεν μπορούν να υποστηριχθούν. Εκείνο όμως το οποίο δεν μπορούμε να δεχθούμε, για παράδειγμα, είναι να ρυθμίζονται θέματα στο επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ δεν ανήκουν σε... Σας ευχαριστώ. Τελευταίες τρεις επεξηγήσεις ψήφου προβλέπεται οι επεξηγήσεις ψήφου να μην μπορούν να ε. παρουσιάζονται μετά την αρχή αλλά εν πάση περιπτώσει κάναμε δυο, ας κάνουμε και άλλες τρεις σε αυτή την περίπτωση οπότε ντόκες για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, αξιότιμε πρόεδρε. Λυπούμε, δεν είχα ζητήσει προηγούμενα να παρέμβω. Η αρνητική αντιμετώπιση μειονοτήτων και ε, ως ε, εμπνεόμενος από θρησκευτικά ιδεώδη πρέπει να πω ότι με την δυνατότητα επίτευξης ενός συμβιβασμού για αυτή την έκθεση για τα θεμελιώδη δικαιώματα υπερψήφισα στο τέλος αυτή την έκθεση του κυρίου Κατάνια. Όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα πιστεύω ότι έχουμε σημειώσει, σημειώνουμε μεγάλες προόδους σε αυτό το πλαίσιο και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για το ότι υπάρχει και το κεφάλαιο για τις που έχει ενταχθεί σε αυτή την έκθεση. Είναι μια απαρχία αυτό ώστε το ένομο σύστημα υπέρ της προστασίας των μειονοτήτων να θεσπιστεί και να λειτουργήσει. Με αυτά τα οποία αναφέρθηκαν προηγούμενα μπορώ να συμφωνήσω. Χρειαζόμαστε ένα συμβιβασμό. Αληθεύει αυτό. Μια και δεν είμαστε σε όλα τα σημεία σύμφωνοι. Για παράδειγμα όσον αφορά τους ομοφιλόφιλους την ευθανασία και συναφή θέματα. Και γι' αυτό δεν μπορώ να δεχτώ οι ηγέτες, θρησκευτικοί ηγέτες να παρεμποδίζονται και να μην μπορούν να δράσουν. Ιδιαίτερα όσον αφορά το σημείο για τους ομοφιλόφιλους. Στην παράγραφο 49 που προαναφέρθηκε, οι παραδοσιακές μειονότητες εδώ και τα κοινοτικά δικαιώματα δεν εντάχθηκαν. Και όσον αφορά και την ατονομία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταψήφισα την έκθεση αυτήν. Παρόλα αυτά μερικές πτυχές της τις υποστηρίζω. Κατεψήφισα διότι στην έκθεση αυτή αναφέρονται μεταξύ των παραδοσιακών μειονοτήτων και οικονομικοί μετανάστες ας πούμε που ήρθαν στη χώρα μου μετά την κατοχή που επιβλήθηκε μετά τον πόλεμο και έτσι Μόνο μισή Λετωνοί μένουν πια στη χώρα μας. Στην ε, πρωτεύουσα τη Ρήγα είναι μειονότητα. Οι ίδιοι οι Λιθουανοί. Ο κύριος Μαντάλταν. Μόλις ψηφίσαμε για την έκθεση Κατάνια και με μεγάλη λύπη εγώ και οι άλλοι δύο Μαλτέζοι συνάδελφοί μου χρειάστηκε να απόσχουμε. Η έκθεση βέβαια αναφέρεται σε πολλά θέματα που ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά περιλαμβάνει και την έκτρωση που δεν έπρεπε να περιλαμβάνεται. Οι Μαλτέζοι εκπρόσωποι στο Κοινοβούλιο είναι κατά των εκτρώσεων και γι' αυτό χρειάστηκε να καταψηφίσουμε το τμήμα αυτό της έκθεσης. Υπάρχουν όμως και άλλα όπως το δικαίωμα μιας αξιο, ενός αξιοπρεπούς τέλους της ζωής επί των οποίων απέσχομεν επίσης και γι' αυτό απέσχομεν και στο τέλος. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Και τώρα πάμε στι επεξηγήσει ψήφου για την έκθεση ΚΑΠΑ. Το ήδη ακούσαμε προηγουμένω τον κύριο Μίτσελ και τώρα η κυρία Ρόιτοβα. Εγώ υποστήριξα αυτό το κείμενο. Ε, δεν, ε, υποστήριξα αυτό το κείμενο που είναι πολύ λαϊκιστικό. Στο αρχικό του κείμενο συμπεριλάμβανε διάφορες θετικές ρήτρες. δυστυχώ δυστυχώς άλλαξε. Ε, εγώ δεν θέλω να υποστηρίξω πράγματα όπως η δημοσίευση εγγράφων τα οποία ανταλλάσσουν μεταξύ τους οι ευρωβουλευτές ή που λαμβάνουν έγγραφα από διάφορες οργανώσεις. Δεν είναι απόρριτα, αλλά εν πάση περιπτώσει καμία ε, συμπολιτισμένη δημοκρατία δεν κάνει κάτι τέτοιο. Τέλος. Ο κύριος Καμάλα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τα πολύ γενικά σας λόγια. Εγώ νομίζω πως όταν μιλάμε για διαφάνεια και πρόσβαση στα ευρωπαϊκά έγγραφα, ε, αυτό είναι κάτι που, επί το οποίο μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε, διότι στο κάτω-κάτω της γραφής είμαστε εδώ, διότι οι φορολογούμενοι είναι αυτοί που μας ψήφισαν και που δημιούργησαν αυτήν τους θεσμούς και χρηματοδοτούν ε, το σώμα και τη δουλειά μας πρόσβαση στα έγγραφα. Να είμαστε βέβαιοι πως ο φορολογούμενος θα έχει πρόσβαση στα έγγραφα που θέλει. Πρόσφατα, μια, η ομάδα των αρχηγών ε, των ομάδων εδώ επισκέφθηκε τη τσεχική δημοκρατία το... και τον αρχηγό της. Αυτός όμως προσέβα... Ε, και μάλλον και ο αρχηγός αυτής της ομάδας προσέβαλε τον πρόεδρο αυτής της χώρας και όλοι ζητούν τη δημοσίευση των πρακτικών εκείνης συνεδρίασης. Ωστόσο, ας είμαστε διαφανείς και ας έχουμε σεβασμό για εκείνους που έχουν διαφορετική άποψη από αυτούς που βρίσκονται εδώ εντός έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι ολοκληρώνονται οι επεξηγήσεις ψήφου. Μπορούμε να σταματήσουμε τις συνεδρίες, θα ξαναρχίσουμε στις 3 με τη συζήτηση για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την Γάζα. Καλή όρεξη σε όλους.